με βάση την ημερήσια διάταξη που καθόρισε η διάσκεψη των Προέδρων 15 Ιανουαρίου. Η ημερήσια αυτή διάταξη έχει διανεμηθεί. Η ομάδα του ΕΛΚ έκανε αίτηση για συζήτηση για τα μέτρα κατά πολέμησης της τρομοκρατίας ζητώντας να υποβληθεί ψήφισμα που θα αποφασιστεί ε, στην πρώτη ολομένη του Φεβρουαρίου. Για να αιτιολογήσει το αίτημα θα μιλήσει ο κύριος Γκονθάλεφ Πόνς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο ε, αποφασίζει επί πολλών ειδών ψηφισμάτων. Μετά τα γεγονότα στο Παρίσι δεν θα είχε καμία έννοια να μην υπάρξει ψήφισμα για το θέμα αυτό η παγκόσμια κοινή γνώμη θέλει να ακούσει τη φωνή της Ευρώπης μέσω του Κοινοβουλίου για την τρομοκρατία. Αλλά επιπλέον και πιο σημαντικό πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε όχι μόνο για να διαδηλώσουμε από κοινού στο Παρίσι, αλλά και επί της ουσίας του θέματος. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η τρομοκρατία, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί απλώς να κάνει συζητήσεις και να μην συμφωνεί επί ψηφίσματος. Γιατί να μην έχουμε ένα ψήφισμα για τον, ε, για την τρομοκρατία θα ήταν η χειρότερη λύση. Γιατί θα απεδείκνει ότι είμαστε μαζί στις διαδηλώσεις, αλλά επί της ουσίας του θέματος δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Είναι απέτηση. Ευχαριστώ κύριε Γκονθάλεθ Πόνς. Θέλει να μιλήσει κανείς υπέρ του ψηφίσματος. Υπέρ παρακαλώ του ψηφίσματος. Ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαίρομαι γιατί ο συνάδελφός μου από το ΕΛΚ θέλει συζήτηση για τις επιθέσεις στο Παρίσι και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Γιατί θυμάμαι κατά τη, ότι κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Προέδρων την προηγούμενη φορά το ΕΛΚ δεν είχε πιστεί ότι πρέπει να γίνει συζήτηση ούτε σήμερα για αυτό το θέμα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για αυτή την αλλαγή στάσης και προτείνω να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση του Κοινοβουλίου πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 του μηνός. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς κατά του ψηφίσματος. Η κυρία Ζήπαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πολίτες έκαναν διαδηλώσεις για τη δημοκρατία, την ελευθερία, για την υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης άποψης και πολλών άλλων αξιών. Χθες η Επιτροπή είπε δεν πρέπει να κάνουμε διάφορες ενέργειες για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και πρέπει να μην καλύψει αυτό το ότι δεν εφαρμόζουμε αυτά που έχουμε ήδη αποφασίσει. αποφασίσει. Ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, ιδιαίτερα την τρομοκρατία που προκύπτει από τις ίδιες μας τις χώρες. Η ριζοσπαστικοποίηση. Οι μαχητές δεν είναι από τρίτες χώρες, είναι πολίτες μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα ήταν άσκοπο έτσι στα γρήγορα να ορνηθοσκαλίσουμε κάτι. Το θέμα είναι να εξετάσουμε όλα τα δυνατά μέτρα και μετά από κοινού να λάβουμε θέση. Γι' αυτό όχι στα γρήγορα απόφαση και ψήφισμα το Φεβρουάριο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ του να υπάρξει ψήφισμα κατά την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά, παρακαλώ. Ωραία, να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λοιπόν, να ξαναρωτήσω, ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας. 205 υπέρ κατά 140 15 αποχές. Η ομάδα των Πρασίνων έχει ζητήσει να γίνει μια συζήτηση για μια δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πάτηση εκπροσώπου για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και της επίθεσης στην Μαριούπολη και προτείνει να συμπεριληφθεί στην ημέρηση διάταξη πριν από τις ε, ομιλίες ενός λεπτού οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 9 η Ολομέλεια για να αιτιολογήσει το αίτημα αυτό η κυρία Χάρμς. Πρόεδρε συνάδελφοι, η ομάδα μου υπέβαλε αυτό το αίτημα και μάλιστα ακόμη και χωρίς την κυρία Μογκερίνη να κάνουμε συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια για τα γεγονότα στη Μαριούπολη και την Ανατολική Ουκρανία. Να παραταθεί κατά μία ώρα δηλαδή Ολομέλεια. Δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε τα ίδια που αποφασίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Υποβάλλουμε αυτό το αίτημα γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ακριβώς μετά από αυτά τα αποτρόπα γεγονότα στην Ανατολική Ουκρανία να καταστήσουμε σαφές ότι τα παρακολουθούμε όλα αυτά, ότι τους αποδίδουμε την αναγκαία σοβαρότητα, ότι και στόχος της πολιτικής μας ε, εργασίας για την Ουκρανία και έναντι της Ρωσίας είναι να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια. Να επανέλθουν. Και η τρομερή καταστροφή και τα δεινά και οι δολοφονίες στην Ανατολική Ουκρανία να σταματήσουν και αποφασίσαμε και μένουμε ότι είναι σωστό να το συζητήσουμε σήμερα γιατί με αγανάκτησαν ε, αυτά που ακούω από διάφορα κράτη-μέλη και ιδίως από την Αθήνα από όπου μας εστάλει το μήνυμα ότι στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλιώς τη Ρωσία σε αυτήν τη σύγκρουση. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναντι του Συμβουλίου των Υπουργών. Αυτή τη βδομάδα, πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών, πρέπει να καταστήσει σαφέ ότι η θέση μα εξακολουθεί να ισχύει και ότι ενιαία και με αλληλεγγύη θέλουμε να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και το Συμβούλιο των Υπουργών και το, η συνάντηση κορυφής. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς λέει. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είναι κανείς άλλος υπέρ του αιτήματο. Θέλει να μιλήσει κανείς υπέρ του αιτήματο, παρακαλώ. Θε... Υπέρ του αιτήματο, όχι. Ωραία. Κατά, ο Σνάλφο Πρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συμφωνούμε με το αίτημα της συναδέλφου γιατί έχει ήδη γίνει μια συζήτηση τη Δευτέρα στην Επιτροπή Εξωτερικών παρουσία και του πρεσβευτού της Ουκρανίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση και του εξηγήσαμε λεπτομερώς τη στάση μας. Δεν έχουμε τίποτε να προσθέσουμε. Αντίθετα συμφωνώ ότι ως προς τη στάση των Αθηνών, διότι όλοι εκπλαγήκαμε όταν μάθαμε αυτή την απαράδεκτη στάση και Πρέπει να το πούμε εδώ ρητά. Είναι απαράδεκτο αυτό που θέλει να κάνει ο Τσίπρας με τον Μπούτιν. Λοιπόν, να ψηφίσουμε επί του αιτήματο. Λοιπόν, να γίνει συζήτηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην ψηφίσετε ακόμη, να ξέρετε γιατί θα ψηφίσετε. Ναι. Είστε πολύ γρήγοροι σήμερα. Να γίνει μια δήλωση. Μπορεί να γίνει από την Κομισιόν ακόμη και αν δεν είναι παρούσα η κυρία Μογκερίνη. Θα είναι μια δήλωση της Κομισιόν. Για την κλιμάκωση τη σύγκρουση στην Ουκρανία και την επίθεση στην, Ουκρανία, στην Μαριούπολη και να συνεχιστεί να παραταθεί η ολομέρεια με τη Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά, παρακαλώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, ήταν σαφές, απορρίπτεται. Όχι, απορρίπτεται. Όχι, δεν χρειάζεται να το ελέγξουμε. Οπότε, καθορίστηκε το πρόγραμμα εργασιών.